για την πράσπιση τη τιμή τη κυρία Κρού. Ενδεχομένω να πρέπει να ληφθούν από κοινού μέτρα. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σα αναφέρω μία περίπτωση η οποία με ανησυχεί ιδιαίτερα και θα πρέπει να μα ανησυχούν όλοι. Πρόκειται για έναν δημοσιογράφο από τη Σιδική Αραβία, Ράμσα Κασγκάρι ονομάζεται. Αυτό ο νέο δημοσιογράφο ε, κατηγορείται για βλασφημία στο λογαριασμό Twitter και κατόπιν αιτήματο τη Σαουδική Αραβία ε, εκδόθηκε στην Σαουδική Αραβία, βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία λόγω των υποτιθέμενων βλασφημιών και απειλείται με εκτέλεση. οι θρησκευτικέ πεπιθήσει ασφαλώ του κάθε ανθρώπου είναι, πρέπει να γίνονται σεβαστέ και αυτό περιορίζει και του δημοσιογράφου. Αλλά η ελευθεροτυπία και η ελευθερία σκέψη είναι ε, καθολικέ αρχέ λόγω ενός ποίηματος του ένας νερός δημοσιογράφος να απειλείται με εκτέλεση στη Σαουδική Αραβία ασφαλώς και δεν, αποδεκτεί, δεν αποτελεί αποδεκτό γεγονός. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε ό,τι περνάμε από το χέρι μας για να αποφευχθεί αυτή η εκτέλεση. Πολλοί συναδελφοί επίσης μου ανέφεραν το γεγονός ότι το Ολλανδικό Κόμμα ΠΕΒΒ δημιούργησε μία ιστοσελίδα στην οποία καλεί να ε, προβληθούν ε, παράπονα για ε, πολίτες Ανατολικής Ευρώπης που κάνουν παραβιάσεις του εργατικού δικαίου. Και η κυρία Ρέντινγκ προέβησε δηλώσεις και διατείνεται ότι πρόκειται για μια ανοιχτή ήπειρος όπου είναι ελεύθερη η μετακίνηση των εργαζομένων. Και μετά από έκκληση πολλών συναδέλφων, χωρίς να γνωρίζω φυσικά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, θα ενημερωθώ για το θέμα αυτό και πρόκειται να συνδυθώ στις αρχές Μαρτίου με τον Πρωθυπουργό Θα το συζητήσουμε το ναι. θέμα αυτό και θα θίξουμε και θα λάβουμε υπόψη και τις ε, ε, ε απόψεις της κυρίας Γκρέτινγκ, η κυρία Βόρτμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχει ανοίξει και ένα site στην Ευρώπη, στην Ολλανδία, για την υποστήριξη της Πολωνίας, όπου όσοι διαφωνούν με την ιστοσελίδα αυτή μπορούν ε, να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους με την Πολωνία. Άρα όλοι οι συνάδελφοι που θέλουν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους μπορούν να το κάνουν σε αυτή την ιστοσελίδα www.propoland.nl Ευχαριστούμε. Ο κύριος Περόν ζητεί το λόγο. Πρόεδρε, Άκουσα την υπεράσπιση της ελευθερίας έκφρασης του δημοσιογράφου της Ειδική αλλά νομίζω πως υπάρχει μια αντίφαση, γιατί νομίζω ότι υπάρχει ε, λόγο, αλλά ε, ε, θέλουμε να υπάρχει ελευθερία έκφραση, θα πρέπει να πούμε το ίδιο και για τον δημοσιογράφο της Ουγγαρίας. Ε, Γενικώ να ισχύει η ελευθερία έκφρασης. Κυρία Σπερώνη, νομίζω ότι δεν με ακούσατε με προσοχή. Ιδάλω δεν θα μπορούσατε να έχετε κάνει αυτή την παρατήρηση. Κυρία Έντφελτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά από αυτά που είπε και η συνάδελφος Βόρτμαν Κόλ, θα ήθελα να πω ότι είναι συμπαθητική ε, φυσικά αυτή η πρωτοβουλία, αλλά νομίζω ότι θα άρμοζε να εκφραστεί δημοσίως το Κοινοβούλιο για την ε, απεχθή αυτή πρωτοβουλία της, ε, του κόμματος ΠΕΒΕΒΕ που καλεί ανώνυμα πολίτες να κάνουν καταγγελίες για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωση και νομίζω ότι θα ήταν προ όφελο τη Ολλανδική κυβέρνηση και θα ήταν προς ε, τη τη να απομακρυνθεί από τα σχόλια αυτά. Yeah, Ο πρόεδρο. κυρία Εντφέλτ, θα πρέπει να σα πω ότι μετά από έκκληση πολλών συναδέλφων ε, αποφάσισα να το κοιτάξω το θέμα αυτό. Δεν το γνωρίζω το, την ιστοσελίδα. Θα έρθω σε επαφή με την κυρία Ρέντινγκ και ενδεχομένω να παρακαλέσω και την Επιτροπή ε, Δικαιώματων, Δικαιωμάτων του Πολίτη να έρθει σε να, να κοιτάξετε την ιστοσελίδα αυτή, αλλά να καλέσω τους συναδέλφους να εκφράσουν την υποστήριξή τους στο website που ανέφερε η κυρία Βόρτμαν Κόλλο. Δεν έχω άλλα τέτοια θέματα στην ημερήσια διάταξη, γι' αυτό να περάσουμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξη. Η κατάσταση των αστέγων στην Ευρώπη λόγω του κύματος